Der Präsident! Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά, συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς και τα εγκεκριμένα κείμενα έχουν διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσει σχετικά. Άλλος θεωρούνται τα συνοπτικά πρακτικά ε, εγκεκριμένα. Ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση για την κατάσταση στη Συρία. Ακολουθεί η δήλωση